τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της σήμερα θα μεταδοθούν ε, ως ε, ήθιστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κέλλη, ευχαριστώ εις το μόνο σας, σας ευχαριστώ